τροποποίησης. Επειδή ακριβώς οι ψηφοφορίες στην Ολομέλεια ξεκινούν 11.30, μειώνεται και κατά ε, μισή ώρα η διάρκεια της δικής μας συνεδρίασης. Ε, τα σημεία 9, 13, 14 αναβάλλονται για την επόμενη συνεδρίαση που θα γίνει 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Για τον ίδιο λόγο θα μειωθεί η συζήτηση για το σημείο 4, τον προπολογισμό του 2018 και για το σημείο 8, δημοσιονομικό, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο κύριος Γκάγιος ζήτησε να συζητηθούν πριν τα σημεία 6 και 7 για το διορθωτικό και για το μέσο ευελιξίας. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τις δύο αυτές εκθέσεις αμέσως μετά τις ψηφοφορίες. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, Θεωρώ ότι μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερησία διάταξη όπως τροποποιήθηκε. Όπως λοιπόν επιθυμούν οι συντονιστές, θα δούμε το πώς προχωρούν διαπραγματεύσεις μεταξύ της Βρετανικής κυβέρνησης και της Ένωσης για το Brexit. Διαπραγματευτής ο Γκίφερ Χόφστατ που θα είναι παρόν στις 10 Οκτωβρίου το πρωί στην Επιτροπή μας. Το ωράριο θα το ξέρουμε αργότερα και ελπίζουμε να είναι παρόντες και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει πολλή πολιτική συμφωνία με το Συμβούλιο από την Τρίτη για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, επιμήκυνση. Και θα κάνουμε τώρα ό,τι μπορούμε για να έχει ολοκληρωθεί το κείμενο ώστε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε το συντομότερο δυνατόν στην Ολομέλεια, ούτω ώστε να μπορεί να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2018. Συγχαρητήρια στον εισηγητή μα, τον κύριο Φερναντέ. Οι συντονιστέ τώρα. Σήμερα το πρωί. Ναι, να το συγχαρητήρια, να μην τον χειροκροτήσουμε. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, συντονιστέ όρισαν τον Hans για ε, την, για την έκθεση για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξία για το Ταμείο Βιώσιμη Ανάπτυξη επιφόρσαν τον πρόεδρο, τον υποφαινόμενο, να αναλάβει την εκπόνηση της έκθεσης για την δημοσιονομική καθάριση για την ΕΚΑΧ, η Γκούε ανέλαβε να ορίσει εισηγητή για την υλοποίηση του χρηματοδοτικού μέσου για τις εξωτερικές δράσεις, ενδιάμεση αναθεώρηση και δημοσιονομικό πολιετές, δημοσιονομικό πέραν του 2020, αρχιτεκτονική του πλαισίου. Αυτά ήθελα να θέσω υπόψη σας. Έχετε λάβει το σχέδιο πρακτικών για τις συνεδρίες 19-20 Ιουνίου και αν δεν έχετε αντιρρήσεις, ε, τα πρακτικά θα εγκριθούν. Και ερχόμαστε στις ψηφοφορίες. Παρακαλώ να βάλτε την κάρτα ψηφοφορία στο μηχάνημα. Δεν έχω την κάρτα μου, ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ. Ποιος δεν έχει κάρτα. Mm -hmm. Δύο, τρεις. Και ο πρόεδρος. Bon, le Λοιπόν, πρώτη ψηφοφορία αφορά την απόφαση 18 γενική έκθεση για την έκθεση του Γιάννη Γκάι. Απόφαση 18. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι ή όχι. Λείπει μία ψήφος. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 23 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, μία αποχή. Ποιοι ήταν αυτοί που θέλαν να ψηφίσουν υπέρ και δεν μπόρεσαν. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Άρα 28 είναι οι ψήφοι υπέρ. Ερχόμαστε τώρα στην έκθεση Τάραντ για τα λοιπά τμήματα του προπολογισμού 2017 μεταφορές πιστώσεων. Α, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση, θεωρούμε ότι εγκρίνονται. Ακόμα καλύτερα, κτίρια. Κύριε Χολμάιρ δεν είναι σήμερα μαζί μας βέβαια. Α, σε έψαχνα εκεί και είσαι εδώ. Εντάξει, συγγνώμη. Να σου δώσω το λόγο. Ähm, Γρήγορα σήμερα κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ λίγο. Πρώτα απ' όλα για το Λίβανο, σκιώδης συγητής και εγώ καθίσαμε και συζητήσαμε για το Λίβανο και για το Νεπάλ. Ε, στο Λίβανο δεν υπήρχαν καθόλου ερωτήσεις, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, είναι αναγκαίο και σημαντικό για όλα τα υπόλοιπα. Μπορείτε να τα βρείτε στην εφαρμογή ή κομίτη. Το θέμα είναι απλά ότι θα πρέπει να έχουν οι συνεργάτες μας λογικές κτηριακές εγκαταστάσεις για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους ε, και βεβαίως ε, το θέμα τώρα του Λιβάνου είναι ιδιαίτερο σημαντικό γιατί έχει αυξηθεί κατά πολύ ο αριθμός των προσφύγων στην χώρα. Δεύτερον, έχουμε το κτίριο στο Νεπάλ. Εκεί πέρα υπήρχαν πολλές ερωτήσεις από τους ε, συναδέλφους και μάλιστα είχαμε και μια συζήτηση κάτι με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μας είπε πως ε, πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί στο Νεπάλ ε, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη στελέχωση και είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν κτίρια στο Κατμαντού γιατί πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν διαθέσιμα και μετά τον τελευταίο σεισμό που ήταν της κλίμακας των 9,8 ε, αντιλαμβάνεστε ότι ε, πρέπει να γίνουν ανακαινήσεις γιατί βρίσκονται σε ένα κτίριο το οποίο έχει κρυθεί κατεδαφιστέο. Οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα όπως αντιλαμβάνεστε, γι' αυτό είναι ακριβό το κόστος το κτηριακό, αλλά ε, ο δεύτερος ε, ε, μειοδότης ε, ήταν 1% είχε διαφορά στην τιμή. Γι' αυτό σας παρακαλώ να υπερψηφίσετε και τα δύο αυτά θέματα. Τα μπορείτε να δείτε ανα πάση στιγμή τα έγγραφα και, και τα δικά μου βεβαίως για να επαληθεύσετε όλους τους αριθμούς οι σκιώδεις ηγητές ε, και εγώ θεωρούμε ε, πάντως ότι πρέπει να εγκριθούν. Και τώρα η διαμαρτυρία μου. Λοιπόν, έχουμε δύο κτίρια της ε, Κομισιόν, μου στέλνουν 20 email συνεχώς ότι πληρώνουμε, πρέπει να πληρώσουμε λιγότερο νίκη για τα ίδια κτίρια. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπαίνει στην ημερήσια διάταξη, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε, Μόνικα. Ο κύριος Δεπρέ. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Επειδή εγώ στην προηγούμενη συνεδρία είχα θέσει το πρόβλημα του κόστου των επενδύσεων ε, στο Νεπάλ, ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Χολμάγερ που διοργάνωσε συνεδρίαση μαζί με την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση για να ενημερωθούμε. Και πρέπει να πω ότι εδώ αναγκαστικά θα δεχτώ το προφανέ ότι δηλαδή η επιλογή ε, έγινε βάσει των επιτακτικών αναγκών για τα κτίρια που πρέπει να επιλεγούν. Ε, ευχαριστώ που ενημερωθήκαμε για την ε, γεωπολιτική στρατηγική, η οποία δικαιολογεί αυτή την επένδυσή μα. Λάβαμε το σχετικό σημείωμα. Δεν θα έλεγα ότι είναι άκρο πιστικό, αλλά τουλάχιστον τα επιχειρήματα δικαιολογούν αυτήν την επένδυση. Θα ακολουθήσω λοιπόν τη γραμμή της κυρίας Χολμάγερ. Ευχαριστούμε κύριο Τζάνι. Απλώς ε, μια γενική ερώτηση κι εγώ. Μια-δυο σκέψεις. Γιατί χρειαζόμαστε αντιπροσωπεία στον Νεπάλ. Εγώ δεν καταλαβαίνω σε τι χρειάζεται αυτό προσωπικό. Νομίζω καλύτερο θα ήταν να μην έχουμε καμία αντιπροσωπεία και θα επιβαρύναμε και λιγότερο τον προπολογισμό μας. Η συζήτηση αυτή έχει ολοκληρωθεί. Όσοι ζήτησαν πληροφορίε τι έλαβαν. Να ψηφίσουμε λοιπόν τώρα ποιοι είναι υπέρ ε, τη έκθεση αυτή για τον Επάλη. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Για το Λίβανο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Γκέγερ για το διευθυντικό προπολογισμό υπαριθμό 5. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι για το ότι ε, κάνατε ε, δεχτήκατε να μπουν τα θέματα αυτά στην ημερήσια διάταξη. Δυστυχώς παράλληλα έχω μια άλλη υποχρέωση. Λοιπόν, το σημείο 5, το υπαριθμό 5, είναι η οικονομοτεχνική εργασία για την ε, πολιτική απόφαση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης, ε, αυτό το οποίο λέμε το Ταμείο για την Αφρική εν ολίγης. Γιατί έχουμε ένα ποσό εγγυήσεων που δίνει την δυνατότητα να πάνε τα λεφτά στα αφρικανικά κράτη για να βελτιωθούν εκεί πέρα οι οικονομικές ε, να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση. Εν ολίγης ε, και πολλής αυτά είναι τα πράγματα. Η εγγύηση είναι αρκετά μεγάλη, 1,7 δισεκατομμύρια. Χαίρομαι ιδιαίτερως για το ότι τα κράτη-μέλη ε, δεν ενέγραψαν το κόστος ολόκληρο στον κοινοτικό προπολογισμό, αλλά 400 εκατομμύρια είναι από το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο και 350 εκατομμύρια παραμένουν στον ε, κοινοτικό προπολογισμό προϋπολογισμό και από αυτά οπωσδήποτε 75 ε, εκατομμύρια σε δόσεις των 25 εκατομμυρίων θα διατηθούν από τον επόμενο προϋπολογισμό, δηλαδή 275 εκατομμύρια από τον επόμενο προϋπολογισμό με τον διορθωτικό προϋπολογισμό υπαριθμών 5. Ο διορθωτικός προϋπολογισμός 5 θα χρηματοδοτηθεί από το μέσο ευελιξίας ε, για να μην ε, υπάρξει μεγάλη αλλαγή στον ε, προϋπολογισμό. Αυτά είχα να πω για το διορθωτικό υπαριθμών 5 και αν μου επιτρέπετε να περάσω και στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης που έχει άμεση σχέση με αυτό αφορά την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας ακριβώς για να διατεθεί αυτό το ποσό. Ταυτόχρονα συμβαίνει και κάτι άλλο στον πέμπτο διορθωτικό προϋπολογισμό. Έχουμε στο πλαίσιο των μεγάλων πολιτικών συμφωνιών που είχαμε τον Νοέμβριο για τον προϋπολογισμό του 2017. Είπαμε το τι θα γίνει με την αναθεώρηση του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού προγραμματισμού. Έχουμε κινητοποιήσει 500 εκατομμύρια ευρώ για την πρωτοβουλία για την νεολαία και κινητοποιούμε τώρα εκ των υστέρων ε, και την ε, αύξηση του αποθεματικού ανάγκης ε, από 280 σε 300 εκατομμύρια όλα αυτά σε τιμές του 2011 δηλαδή σήμερα μιλάμε για μια κινητοποίηση 22,8 εκατομμυρίων ευρώ. Τα νούμερα για το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης ε, και Ένταξης ε, περιακόπησαν ε, σημαντικά. Όπως βλέπετε έχουμε λοιπόν την εφαρμογή των έργων του, που θα πληρωθούν από αυτό το Ταμείο γιατί τα έργα υλοποιούνται στα κράτη-μέλη αργότερα από όσο περιμέναμε. Τα κράτη-μέλη μόλις την Άνοιξη φέτος έστειλαν τα ποσά και τις αρμόδιες αρχές που θα ασχοληθούν με αυτά. Οπότε δεν θα μπορέσουν να ρεύσουν πλήρως τα ποσά το 2017, οπότε μπορούμε να μεταφέρουμε λεφτά από εκεί και το έχουμε ήδη συζητήσει στη συνεδρίαση των ε, συντονιστών. Ε, και εδώ πέρα βεβαίως συμφωνώ με τα επιχειρήματα του Ζίγκφριντ Μουρεσάν, ότι δηλαδή εάν ε, τα κράτη-μέλη ζητήσουν κατεπηγόντως κονδύλια για αυτό το ταμείο, τότε ε, ίσως να μην είναι τόσο κατεπήγον το ζήτημα όσο μας λέει το Συμβούλιο και μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε κάποια άλλα πράγματα από αυτό. Merci. Ευχαριστούμε κύριε Γενική Εισηγητά. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Όχι. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι θα είστε στο Συμβούλιο για το Διευθυντικό 5 στις 28 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι λίγη η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών Στις 10 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Προπολογισμών και στην Ολομέλεια 23 ή 26 Οκτωβρίου. Υπαριθμών 7 πάλι ο κύριος Γκάγερ διοργάνωση των ε, μέσων ευελιξία. Αναβάλλετε. Ε, το είπα. Μόλις το είπα, κύριε Πρόεδρε. καλοντριέ. Ε, Α, ίδιο χρονοδιάγραμμα λοιπόν. Η κυρία Βάιντερ θέλει τώρα το λόγο νομίζω γιατί έχει αντιμένες υποχρεώσει. Παρακαλώ. Si le rapporteur général Συμφωνείτε κύριε Γενική Εισηγητά. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το Ταμείο Αλληλεγγύης ε, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση μιζώνων ε, καταστροφών και θέλουμε με τον τρόπο αυτό να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας ε, σε πληγές περιοχές Ευρώπης. 500 ε, εκατομμύρια είναι το ανώτατο όριο κατέτος με τιμές 2011 πάνω από τις κατηγορίες σχετικού πλαισίου. Ο στόχος της σχεδίου έκθεσης που είναι εκ των προτέρων να έχουμε τις αναλήψεις υποχρεώσεων για τον προϋπολισμό του 2018. Η πληρωμή προκαταβολών θα μας δώσουν τη δυνατότητα να αντιδρούμε έγκαιρα, αποτελεσματικά σε περίπτωση καταστροφής. Το 2018 το συνολικό ποσό των προκατάβολων ήταν 5 εκατομμύρια στις αναλήψεις και στις υποχρεώσεις και στις πληρωμές. Σε ό,τι αφορά τις προκαταβολές, το ποσό δεν πρέπει να υπερβαίνει, όπως γνωρίζουμε, το 10% των χρηματοδοτικών εισφορών που μπορούμε να προβλέψουμε. Το Ταμείο Αλληλεγγύης, για να υπογραμμίσω, δεν είναι ένα απλό χρηματοδοτικό μέσο, είναι μια πλατφόρμα αλληλεγγύης, είναι ένα όχημα μέσω των οποίων μπορούμε να εκπέμψουμε ηχηρά πολιτικά μηνύματα προς τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πληγεί από κάποια καταστροφή. Χθε εγκρίθηκε η μεγαλύτερη δυνατή κινητοποίηση, μάλλον μεγαλύτερη κινητοποίηση μέχρι τώρα του Ταμείου Ελληνικής 1,2 δις χρηματοδοτική βοήθεια στην Ιταλία. Κατόπιν τούτου, το 2018 ξεκινάμε χωρίς ε, πλεόνασμα χρηματοδότηση από τα προηγούμενα χρόνια σε αυτό το ταμείο. Γι' αυτό λοιπόν Ελπίζουμε να μας δείξει έλεος η φύση στο μέλλον. Μίλησα για τις προηγούμενες προκαταβολές, ε, τον προκλήσιμο του 2018. Ελπίζω να συμφωνείτε με αυτά που είπα. Ευχαριστούμε πολύ. Παρατηρήσεις υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Το χρονοδιάγραμμα το ίδιο και για το γενικό προπολογισμό για την υποβολή τροπολογιών, την ψηφοφορία στην Επιτροπή μας και την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Οπότε περνάμε στον ε, γενικό εισηγητή, τον κύριο Μούρισαν, για να μας μιλήσει για τον προϋπολογισμό ε, του 2018, την κατάρτιση, πώς ε, βλέπετε τις πολλές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, θετικά, αρνητικά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τώρα βρισκόμαστε στην φάση την εξής ε, την προηγούμενη εβδομάδα. Όλες οι τροπολογίες ε, κατατέθηκαν. Πριν από δύο εβδομάδες ήταν στις επιτροπές και την προηγούμενη εβδομάδα ήταν οι πολιτικές ομάδες. Οπότε την ε, προηγούμενη Παρασκευή μαζί με την γραμματεία της Επιτροπής Προπολογισμού, την οποία οφείλω να ευχαριστήσω, κάναμε μια προσωμείωση του τι μπορούμε να κάνουμε με τους περιορισμένους πόρους μας. Και αυτή την εβδομάδα, σε μόνιμη επαφή με τους σκιώδεις εισηγητές, κύριε Πρόεδρε, για να καταρτήσουμε ένα συμβιβαστικό πακέτο, το οποίο θα ψηφιστεί μετά την πράσινη εβδομάδα στην Επιτροπή Προπολογισμών στις Βρυξέλλες και μετά στην Ολομέλεια στο τέλος Οκτωβρίου. Ο στόχος είναι να έχουμε μια ξεκάθαρη θέση για τις ε, διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ε, τα αιτήματά μας πρέπει να είναι ρεαλιστικά, λογικά και να γίνουν στις ε, γραμμές όπου υπάρχει όντως ανάγκη για επιπρόσθετη χρηματοδότηση και η πλειοψηφία την οποία σκοπεύω να επιτύχω είναι μεγάλη και γι' αυτό ακριβώς συναντήθηκα με τους κοιόδης ηγητές γιατί χρειαζόμαστε μεγάλη πλειοψηφία για τι διαπραγματεύσει με το Συμβουλίο. Όπω ξέρετε το Συμβουλίο έχει κάνει περικοπές ε, κάποιες από τι οποίε είναι ανεύθυνες για τομεί που επηρεάζουν το μελλοντικό, μελλοντική δύναμη της Ένωσης, έρευνα, καινοτομία, υποδομές και θα ε, ε, αντιταχθούμε στην διαπραγμάτευση, δεν θα τις ε, δεχτούμε. Τώρα λοιπόν είμαστε στη διαδικασία τη συμβαστική. Τι μορφή θα έχει. Πρώτα απ' όλα στον τίτλο 1α έχουμε πολύ περιορισμένο περιθώριο 56 εκατομμύρια ευρώ και το χρησιμοποιούμε αυτό για να ενισχύσουμε ακριβώς τις γραμμές εκείνες που γνωρίζουμε ότι έχουν μεγάλη ζήτηση. Μικρόμεσαίες επιχειρήσει, έρευνα, καινοτομία. Δηλαδή κόσμε, Εράσμους, Μαρή ε, Κιουρί, το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Συμβουλίου και προγράμματα κλιματικής αλλαγής. Ε, βλέπετε ότι το κλίμα όπου είναι δυνατόν έχω προσπαθήσει να το εφαρμόσω. Επίσης έχουμε ζητήσει να αποκαταστήσουμε τις ε, περικοπές στο ΕΦΣΥ. Ένα Β θα ενισχύσουμε την πρωτοβουλία για την νεολαία. Αυτή τη στιγμή κοιτάμε ποιο θα πρέπει να είναι το ακριβές ποσό. Διαφορετικές ομάδες έχουν καταθέσει διαφορετικά ποσά. Τίτλος 2, όπως ξέρετε, στη Γεωργία έχουμε μικρά περιθώρια ελιγμών. Μικρότερα από ό,τι σε άλλους τίτλους. Εδώ πέρα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να αντιδράσουμε σε ε, απρόσμενες ε, κρίσεις. Γι' αυτό το 350 εκατομμύρια ευρώ το περιθώριο θα μείνει άθικτο για πιθανές ε, κρίσεις. Γύρω στα 100, ευρώ θα, 100 εκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτήσουμε για έργα που λένε οι συνάλφοι ότι χρειάζονται και θέλω να δοθεί περισσότερη στήριξη στους νέους αγρότες, γιατί έτσι δημιουργούνται θέσεις εργασίας, θα μειωθεί η ανεργία των νέων στην Ήπεθρο. Τίτλος 3, ε, εκεί πέρα έχουμε λίγα περιθώριο, μηδενικό περιθώριο, αλλά έχουμε το θέμα της βελτίωσης της ασφάλειας ε, των πολιτών, θα ενισχύσουμε τις ε, υπηρεσίες της Ένωσης που έχουν σχετικές αρμοδιότητες, ΕΑΖΟ, Europol, Eurojust, SEPOL, και τίτλος 4 ε, υπήρχε εδώ πέρα το περιθώριο των 250 εκατομμυρίων, 230 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά πρέπει να ξέρουμε αν επεκτείνουμε το μέσο προσφύγων για την Τουρκία πρέπει να αλλάξει λόγος 4. Αλλά μέχρι να ακούσουμε κάτι τέτοιο λειτουργούμε με το πλαίσιο που έχουμε. Δηλαδή να χρησιμοποιηθεί το περιθώριο για να ενισχυθεί η γειτονιά μας και ειδικά η νότια γειτονία. Από εκεί προέρχονται οι προκλήσεις. Γιατί βλέπουμε επίσης και τη Ρωσία που κινητοποιείται. Υπάρχουν χώρες που συνεργάζονται περισσότερο με την Ευρώπη. Ρωσία, Ουκρανία και κοιτάμε και το τι έχουν καταθέσει και οι συνάδελφοι ε, της ε, Επιτροπής Εξωτερικών ε, για το θέμα αυτό και για την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Τουρκία. Προτείνει στην συνάδελφοι να κόψουμε κάποια κονδύλια από την Τουρκία και να μπουν στο αποθεματικό υπό όρους. Δηλαδή να υπάρχει αίρεσιμότητα ε, με όρους την πρόοδο στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εν ολίγης, κύριε Πρόεδρε, αυτά είναι τα θέματα πάνω στα οποία εργαζόμαστε με τους χειοδησηγητές. Τα πιλωτικά και τις προπαρασκευαστικές δράσεις θα προετοιμάσουμε ένα πακέτο για τα πιλωτικά έργα και έχουμε καλές αξιολογήσεις ε, ανάλογα αν το θα έχουμε καλές αξιολογήσεις α ή β. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τις ε, προτεραιότητες που έθεσε το Κοινοβούλιο. Το μήνυμά μου προς όλους τους συναδέλφους είναι να στηρίξουν ε, τις αλλαγές. Ε, πάντα να ξέρετε ότι η πόρτα μου είναι ανοιχτή για να συζητήσουμε τυχόν τροπολογίες και την Πράσινη Εβδομάδα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μουρεσάν για την τόσο πολύτιμη δουλειά σας. Προσπαθήσατε να συνδυάσετε όλες τις πρωτοκίες, ιδίως όλων όσοι έχουν την πρόθεση να ε, ε, δουν και να εγκρίνουν τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018. Κύριε Σασκορθίτη για την πολύ του προπολογισμού, ευχαριστώ, Πρόεδρε να θυμίσω στους συναδέλφους ότι τον Απρίλιο φέτος το Κοινοβούλιο ενέκρινε τον δικό του προπολογισμό. Και να σας θυμίσω ότι αποφασίσαμε άξι 2,3% σε αυτή τη φάση. Με το ποσοστό πληθωρισμού που είχαμε τότε, θεώρησα ότι είναι και δικαιολογημένη και υπεύθυνη στάση. Θέλω λοιπόν να σα στήσω στην Επιτροπή μα και στο Κοινοβούλιο το επίπεδο της αύξησης αυτής 2,3% να θεωρηθεί ως ε, δείκτης αξιολόγησης και για τις υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Με την έκθεση αυτή θα δούμε κατά πόσον, μάλλον δέχτηκαν τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα περίπου αυτή την πρόταση και έχουν παρόμοιε προτάσει. Υπάρχουν τρει εξαιρέσει, ωστόσο, που θα έπρεπε να αναφέρω εδώ στην Επιτροπή. Η πρώτη είναι ο, επόπτης, ο Ευρωπαίος Επόπτης ε, Προσωπικών Δεδομένων. Βρίσκεται ακόμα στα πρώτα βήματα της λειτουργίας του οργανισμός αυτός. Χρειάστηκε να ε, σχηματιστεί νέο διοικητικό συμβούλιο. Οπότε φέτος θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν αυτές τις δραστηριότητες και θα χρειαστεί μία αύξηση του 27,9%. Ξεκίνησε από πολύ, πολύ χαμηλή βάση όμως και είναι στα πρώτα στάδια λειτουργίας της. Δέχομαι λοιπόν αυτόν τον αριθμό ως δικαιολογημένο. Έπειτα το ελεκτικό συνέδριο έχει μια μεγάλη αύξηση στον όγκο εργασιών του. Δέχομαι και εκεί λοιπόν το αίτημά του που είναι δικαιολογημένο και σωστό και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ζήτησε επίση αύξηση στη χρηματοδότηση και εκείνοι γιατί έχουν αντωνότερη δραστηριότητα αλλά και επειδή είχαν κάποια θέματα ασφαλείας προτείνουν αύξηση 2,96% σε σχέση με πέρσι. Δεδομένου ότι υπάρχει αυτό το επιπλέον κόστος, θεωρώ ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να ξανασκεφτεί τις περικοπές που έχει κάνει σε κάποια τα κονδύλια, ε, γιατί είναι προπολικές. Θα πρέπει να επαναφέρουμε ε, στα επίπεδά του κάποια από τα ποσά αυτά πριν τις περικοπές. Ωστόσο, εάν θέλουμε το συνολικό όγκο, τον να τον τηρήσουμε υπό έλεγχο στα πλαίσια του 2,3% συνολικά, θα πρέπει να κάνουμε περαιτέρω εξοικονομήσει. Γι' αυτό λοιπόν θα μπορούσαμε να έχουμε κέρδος ως προς την αποδοτικότητα. Με χαρά αναφέρω εδώ ότι είχαμε επαφές με το ελεκτικό συνέδριο, οι οποίοι σε επιστολή τους προτείνουν να γίνει πρόσθετη περικοπή 750 ε, εκατομμύρια ευρώ περίπου και ότι αυτό μπορεί να γίνει εντός του προβλεπόμενου ως τώρα προπολογισμού. Το άλλο μέρος των περικοπών μας μπορεί να γίνει με ανακατανομή κάποιων χρηματοδοτήσεων. Προς αυτό το σκοπό εξέτασα πολύ ε, προσεκτικά όλα τα κεφάλαια, ιδίως ό,τι αφορά την ΕΟΚΕ, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ε, η οποία έχει προπολογισμό 123 εκατομμύρια ευρώ και την Επιτροπή των Περιφερειών που έχει προπολογισμό 3 εκατομμύρια ευρώ για τη φετινή χρονιά, ε, για το 2018, προτείνω και για του δύο αυτού οργανισμού ένα πάγωμα στον προπολογισμό του. Επίση, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση έχει διαρκώ αυξανόμενο κόστο. Και λόγω τη τελέχωσή τη, εν μέρη, και λόγω τη στατηγική επικοινωνιακή του πολιτική, η οποία εγκρίθηκε και από τι δικέ μα κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Το περισσότερο από αυτό το κόστο μπορεί να απορροφηθεί από, την ΕΕΔ, από τον τρέχοντα προπολογισμό του. Δέχομαι όμω να γίνει μια μικρή προσαρμογή κάποιων εκατομμυρίων ευρώ, ιδίω για να αντιμετωπίσουν τι τρέχουσε ανάγκε του. Το δέχομαι αυτό. Επιπλέον, μετά από συνάντηση με τους κοιότητες εισηγητές την αρχή της εβδομάδας, δέχτηκα και τις δικές τους μέρημνες και άκουσα τα επιχειρήματά τους σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δέχομαι λοιπόν ότι χρειάζονται πρόσθετα κονδύλια λόγω των μεταφραστικών αναγκών και της διερμηνίας. και δέχτηκα 1,9 εκατομμύρια ευρώ να αποδοθεί στον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Για την ΕΕΔ έχω λιγότερη συμπάθεια διότι ο Ευρωπαϊκός Διαμεσολαβητής ζήτησε περισσότερη μαθητεία και άσκηση με 100 εκατομμύρια με 100.000 ευρώ μάλλον επιπλέον. Όμω, παρά τι παραχωρήσει αυτέ ε, στη συνάντηση των σχεδόν, παραμένω απογοητευμένο δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε κοινό έδαφο ε, συνεννόηση για δύο ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, όπω είπα, το ελεγκτικό συνέδριο μα απίφθινε επιστολή όπου προτείνει η περικοπή 750 εκατομμύρια ευρώ, την οποία είπε ότι μπορούσε να δεχτεί. Πραγματικά λοιπόν ξαφνιάζομαι και δεν καταλαβαίνω γιατί οι δύο μεγάλε ομάδε επιμένουν να παραμένουμε στην αρχική χρηματοδότηση του ελεκτικού συνεδρίου. Επιπλέον, παρομοίω για την Επιτροπή των Περιφερειών και την ΕΟΚΕ, δεν πείθομαι από τα επιχειρήματα για αύξηση στη δική τους, ε, στο δικό του προπολογισμό. Εν τέλει, Πρόεδρε, θέλω να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι αν επιθυμούμε να παραμείνουμε κάπου κοντά στον δείκτη συγκριτική αξιολόγηση στο όριο του 2,3% που εμεί οι ίδιοι θέσαμε στον εαυτό μα. Εάν θέλουμε να είναι υπεύθυνη και λογική η αύξηση που θα προτείνουμε, πρέπει να λάβουμε κάποιε σκληρέ αποφάσει. Γι' αυτό θα, θα παρότρινα ε, εντόνω του συναδέλφου να δεχτούν τι συμβαστικέ που του προτείνω. Ευχαριστώ. Merci, Σας ευχαριστούμε, κύριε Άσχουερτ για την παρουσίαση αυτή. που ζητεί κάποια αυστηρότητα και δείχνει όμως και την ε, θέληση για δικαιοσύνη. Από τους κύριους ηγητές ο κύριος Βιώτη. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ να συγχαρώ τις ε, παρατηρήσεις που απευθύνατε και τα συγχαρητήρια στον εισηγητή του Γενικού Προπολογισμού για την προσπάθειά του Πρέπει να δώσουμε μια απάντηση στην τελική του έκκληση. Στηρίζουμε την ανάγκη να έχουμε ένα κοινοβούλιο ενωμένο στη θέση του όταν θα πρέπει να τοποθετηθούμε γενικώ για τον γενικό προπολογισμό. το να παραμένουμε ανοιχτό μυαλί μας επιτρέπει να διαπραγματευόμαστε με κάποια διαλλακτικότητα. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω. Θα ψηφίσουμε όμως την Επιτροπή για να προκύψει η θέση μας και οι διαφωνίες μας δεν είναι και πολλές αριθμητικά, αλλά έχουν πολιτική αξία με κάποια βαρύτητα. Νομίζω όλοι μπορούμε να κατανοήσουμε, παρόλο που έχουμε διαφορετικές θέσεις, όλοι μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν θέσεις για, με διαφορετικές απόψεις για την Ευρώπη που επιθυμεί το Κοινοβούλιο και όχι τόσο πολύ στην κατεύθυνση που επιθυμεί το Συμβούλιο. Τα προβλήματα τα γνωρίζουμε. Η δουλειά που έγινε για το κεφάλαιο 1α και 1-2 για τους τίτλους 1α και 1-2 είναι σημαντική. Προσπαθούμε να ανακτήσουμε τις βασικές περικοπές που είχαν γίνει ιδίω για το ΣΕΦ για το 2020 για το Εράσμους όλα αυτά τα εκτιμούμε και συνδυάζονται και με τις δικές μας πολιτικές θέσεις και με τη γενικότερη θέση του Κοινοβουλίου. Παραμένουν κάποιες σημαντικές διαφορές ως προς την προσέγγιση που θα ακολουθήσουμε για την πρωτοβουλία των νέων. Και εδώ πρέπει να απευθύνω αμέσως μια έκκληση ε, να είμαστε πολύ περισσότερο φιλόδοξοι πρέπει. Το άκουσα σε προηγούμενη συνεδρίαση, κάποιος το είπε, ο συνάδελφος Φερνάντες αναφέρθηκε στην ανάγκη να προτείνουμε λύσεις στους νέους, να είμαστε κοντά τους. Θα πρέπει να σχεδιάσουμε ένα σύστημα όπου θα επενδύσουμε τα δισεκατομμύρια ευρώ που προβλέπουμε για την κινητικότητα των νέων, ναι μεν, αλλά θα πρέπει να γίνουν και τεράστιες προσπάθειες για να κάνουμε κάτι για την απασχόληση των νέων. Επ' αυτού πρέπει να γίνει μια προσπάθεια μεγαλύτερη. Διότι το πρόβλημα είναι η ενεργεία των νέων. Η απασχόλησή τους, που δεν αφορά απλώς λίγες μόνο χώρες, αλλά διατρέχει ολόκληρη την Ευρώπη και την επικράτειά της. Για τις υπόλοιπες γραμμές και πολύ συνοπτικά νομίζω πρέπει να γίνει και άλλη δουλειά εμβάθυνσης για τα θέματα του πολιτισμού και της παιδείας διότι θα χρειαστούμε περιθώρια ιδίως για την επόμενη χρονιά που έχει συγκεκριμένο τίτλο ως έτος. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν συγκεκριμένες προσπάθειες για τον πολιτισμό και όπως έχω πει και άλλες φορές στον τίτλο 4 παραμένουν κάποια προβλήματα. Προβλήματα που πρέπει να τα εξετάσουμε. Απέχουμε από το να έχουμε μια κοινή θεώρηση. Όχι πάρα πολύ, αλλά απέχουμε. Τελευταία μου αναφορά στα πιλωτικά προγράμματα. Και εδώ είναι γνωστή η θέση μας. και τα είχαμε δει και σε συνεδριάσει τη Επιτροπή μα όταν συζητούσαμε τα πιλωτικά προγράμματα και τι προπαρασκευαστικέ δράσει, προτείνω να ακολουθήσουμε μία μέθοδο που να μην είναι απλώς αυτή της ψήφισης και της έγκρισης των πιλωτικών προγραμμάτων, όπως έχει ήδη γίνει από την Επιτροπή μας, αλλά να ακολουθήσουμε ένα κριτήριο που να συνδυάζει ε, και τις πολιτικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου. Δηλαδή, όταν διαλέγουμε το σύνολο των πιλωτικών προγραμμάτων και των προπασκευαστικών ε, δράσεων, ε, εγώ με μια μικρή μου συμβολή και τροπολογία προς τον ε, εισηγητή θα προτείνω να ακολουθούμε όχι μόνο τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, αλλά και τις πολιτικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου μας. Διότι είναι χρέος μας για λόγους ανεξαρτησίας του δικού μας τεχνικού οργάνου να κοιτάξουμε κατά πόσο να ανταποκρινόμαστε και στις ανάγκες των πολιτών που κάτι περιμένουν από εμά και από τον ερχόμενο προπολογισμό. Περιμένουν κάποιες σοβαρές απαντήσεις σε προβλήματά τους. Ευχαριστώ για την ως τώρα συνεργασία. Ο εισηγητή μα είπε ότι ακόμα είναι διαθέσιμο για να συζητήσουμε. Θα εκμεταλλευτώ λοιπόν την ευκαιρία και την ερχόμενη εβδομάδα. Με συγχωρείτε, Πρόεδρε, που δεν μπορούσα να παρακολουθήσω όλη, όλη τη συζήτηση, αλλά ψήφισατε, ψηφίσαμε νωρίτερα και έπρεπε να λείψω. Αφού είστε όμως ακόμα εδώ κύριε Βιώτη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτά που είπατε. Σίγουρα η απασχόληση των νέων είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι σκάνδαλο να υπάρχει τόσο υψηλή νεανική ενεργεία, ιδίω σε μια χώρα που ένα στου δύο νέου είναι άνεργοι. Αλλά χρειάζεται και επαγγελματική κατάρτιση γιατί αυτό επηρεάζει την ε, πρόσβαση στην απασχόληση. Ο κύριος Κέλμελ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Ευχαριστώ και εγώ τον ε, Ρίτσαρντ Άσχουρτ για τη δουλειά που έκανε. Πάρα πολύ δύσκολη και συμφωνώ πλήρως με τα όσα προτείνει και στηρίζω τη γραμμή του. Ε, Πολύ καλά. Να και μία περιεκτική και σαφέστατη παρέμβαση. Κύριε Τάραντ. Ε, Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά την έκθεση του κύριου Μούρεσαν, θα επαναλάβω αυτό που είπα στην των συντονιστών. Και μην πάμε στι πράσινε τροπολογίε γιατί νομίζω λαμβάνονται υπόψη καλά στις συμβαστικές προτάσεις. Συγχαρητήρια λοιπόν και ελπίζω να έχετε αέρα στα πανιά σας στις διαπραγματεύσεις. Για την έκθεση για τα λοιπά τμήματα αναλαμβάνω αυτό που είπε ο κύριος Κέρμελ. Πολύ καλά τα κάνατε κύριε Άσφορντ. Συγχαρητήρια. Merci. Σας ευχαριστώ. Βάλει Ζόλτεκ Φερνάντε, για την άποψη του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω όμως πορτογαλικά, μου επιτρέπετε. Ευχαριστίες και συγχαρητήρια στον εισηγητή για τη δουλειά του, για την φιλοδοξία με την οποία εξέτασε όλες τις προτάσεις και το ρεαλισμό με τον οποίο αντιμετωπίσαμε όλα τα θέματα στη δουλειά όλων των πολιτικών ομάδων ίσχυσε αυτό, όλων των σκηριωδών εισηγητών. Το Κοινοβούλιο ως συνήθως φάνηκε ενωμένο στα θέματα του προπολογισμού. Έχουμε κοινέ προτεραιότητες, ακόμα και αν υπάρχουν διαφορετικές θεωρήσεις για κάποια θέματα. Όλοι θέλουμε την αύξηση, την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι θέλουμε να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, ιδίως για τους νέους. Θεωρούμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι σημαντικές για να επιδιώξουμε αυτό το στόχο. Η καινοτομία και η έρευνα είναι καθοριστική σημασία. Υπό αυτήν την έννοια είναι απαράδεκτο, απίστευτο και ακατανόητο το Συμβούλιο να προτείνει 490, 490 εκατομμύρια ευρώ περικοπές και να θέλει να επιτύχει τους στόχους το 2020. Είναι θλιβερό και αντιφάσκει και με τις ίδιες προτάσεις του Συμβουλίου. Επίσης, απαράδεκτο, είναι η πολιτική συνοχής που είναι καθοριστική σημασία για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ίδια την ανάπτυξη της Ένωσης αλλά και την κοινωνική και πολιτική και οικονομική συνοχή της Ένωσης να περικόπτεται με 200 εκατομμύρια ευρώ ε, να έχει μια τέτοια περικοπή στον προπολογισμό τη. Ε, είναι ακατανόητο κι αυτό. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθήσουμε την απασχόληση, αλλά πολλά εξαρτώνται από τις πρωτοβουλίες των κατών μελών και τη δική μας προσπάθεια να πετύχουμε αυτό το στόχο. ό,τι αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, την εκπαίδευση, και αυτό είναι ζωτική σημασία, αλλά πρέπει να προωθήσουμε την κινητικότητα. Γιατί ε, θα πρέπει να δώσουμε στους πολίτες την αίσθηση ότι η ιδιότητα του ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποιο νόημα. Ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηριχθεί από τι πολιτικέ ομάδε που θέλουν να διατηρηθεί αυτό το εγχείρημα υπεράσπιση τη ειρήνη, των αξιών, τη οικονομική ανάπτυξη και ποιότητα διαβίωση για του πολίτε μα. Και θυμίζω κάτι που πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε, ότι ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και αν είναι 1% του ΑΕΠ, του χώριου προϊόντος για να το πω ακριβέστερα, είναι πολύ απαραίτητο για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε πολλές κρίσεις και πολλά προβλήματα σε πολλές χώρες όπως η Πορτογαλία λόγω χάρη. Ο προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 70% των δημόσιων επενδύσεων. Στην ουσία Μιλάμε για το 90% του προπολογισμού της Ένωσης, κύριε Μουρεσάν. Διοικητικέ δαπάνες είναι ένα κομμάτι, αλλά προϋπολογισμός της Ένωσης κατά 94% αφορά την έρευνα. Είναι πολύ μικρό το κομμάτι που αφορά τη χρηματοδότηση και τις διοικητικέ δαπάνες. Σε αυτό το 94% λοιπόν πρέπει να αποδώσουμε απαραίτητο χρόνο και προσπάθεια. Είναι σημαντικό και το 6% βεβαίω και αυτό χρειάζεται προσοχή γιατί χρειάζεται κάτι ελάχιστο για τη λειτουργία. Αλλά αυτό το ελάχιστο της λειτουργίας ε, απαιτεί να κάνουμε μια τεράστια δουλειά για να ε, επιδιώκει τους στόχους των προπολογισμών και να τους ε, πετυχαίνει. Ευχαριστώ πολύ και τον Ρίτσαρτ Άσχορ για τη δουλειά του στο θέμα αυτό. Συμφωνούμε όλοι ότι ο προπολογισμό των θεσμικών οργάνων, ακόμη και ένα 6% του συνόλου του προπολογισμού, πρέπει να εκτελείται αυστηρά, πρέπει να υπάρχουν οικονομίε συστηματικά, αλλά να δίνει και αρκετού πόρου ώστε να λειτουργούν εύρυθμα τα θεσμικά όργανα. Πρέπει να επιδιώκονται σωστέ προτεραιότητε ε, και να υπάρχει απόκριση στι προκλήσει που έχουμε μπροστά μα. Ελπίζω το Συμβούλιο να έχει την ίδια επικοδομητική στάση διότι πολύ συχνά κάνει περικοπές, αλλά ούτε εξηγεί ούτε δικαιολογεί τα αίτια αυτών των περικοπών, που μπορεί να είναι τελείως αφαίρετες. Γι' αυτό θα ευχηθούμε καλή συνέχεια στον εισηγητή και στην πρότασή του, γιατί έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και είμαι βέβαιο ότι το Κοινοβούλιο θα φανεί ενωμένο για να επιτύχουμε τον κοινό μα στόχο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Φερνάντε που μα εκφράσετε τη θέση τη ομάδα σα, του ΕΛΚ. Για τα υπόλοιπα τμήματα, ο κύριος Ντουσάντος είναι μαζί μας, θέλει να πει τη γνώμη του για τα υπόλοιπα τμήματα. Πρόεδρε, δεν έχω πολλά να προσθέσω. Όντω πρέπει να επενέσω τον εισηγητή Άσκορφ για τη δουλειά του. Ήταν πολύ θετικό στη στάση του. Είχαμε εντατικό διάλογο μεταξύ μα. απλώς σε αυτή τη φάση να πω ότι έχουμε κάποιες μικρές διαφωνίες από την ομάδα μας, ιδίω σε ό,τι αφορά το ελεγκτικό συνέδριο, κάτι που θα διευκρινιστεί στο επόμενο διάστημα, καθώς θα συζητήσουμε απευθείας με το ελεγκτικό συνέδριο και τους εκπροσώπους του και έπειτα μια διαφωνία για τη σημασία που, έχει κάθε, που αποδίδει κάθε πολιτική ομάδα ή κάθε βουλευτή στην Επιτροπή των Περιφερειών. Εγώ θεωρώ ότι η ομάδα μου, οι Σοσιαλιστέ και οι Δημοκράτε, ε, έχει κάποιε πολιτικέ μέρημνε πολύ σαφεί. Ο προπολογισμό είναι ένα εργαλείο πολιτικού χαρακτήρα. Και το είπε μόλι τώρα και ο αγαπημένο μου φίλο ο Φερνάντε. Το είπε και πρόσφατα το Κοινοβούλιο σε τοποθέτησή του. Δεν μπορούμε λοιπόν να κλείσουμε τα μάτια μπροστά σε την πραγματικότητα. Χρειάζεται ορθολογισμός στην επιλογή και την απόδοση των προποδοτήσεων. Όμως, δεν θα πρέπει σε αυτή την προσπάθεια να διακυβεύσουμε την εύρυθμη, να, να θέσουμε ένα την εύρυθμη λειτουργία αλλά και διαφανή λειτουργία κάποιου θεσμικού οργάνου. Ο προπολογισμό αυτό είναι σχετικά μικρό στο σύνολο των όσων συζητούμε. Όμω προφανώς είναι πολύ σημαντικό για το καθένα θεσμικό όργανο ξεχωριστά για να μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει απαραίτητη αξιολόγηση και η απαραίτητη πολιτική αξία στη δουλειά του κάθε θεσμικού οργάνου. Θα κάνουμε λοιπόν τις ανάλογες προσπάθειες από την πλευρά της ομάδας των σοσιαλιστών και δημοκρατών ελπίζοντας ότι στο Συμβούλιο θα γίνει δεκτή η δουλειά του κυρίου Άσφορντ, του εισηγητή μας που είναι πολύ καλή και ε, γιατί οι περισσότερες απόψεις ε, αντικατοπτρίστηκαν στην τελική εκδοχή της πρότασης και αυτό το θεωρούμε πολύ θετικό. Οπότε σκοπεύουμε να ταχθούμε υπέρ της πρότασης αυτής. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Ντουσάντους. Ακούσαμε όλους τους σκιώδεις εισηγητές. Ο γενικός μας εισηγητής θα μπορούσε ενδεχομένως με λίγα λόγια να ολοκληρώσει αυτήν την συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, θα μας βοηθήσουν τα σχόλια τις επόμενες εβδομάδες. Θα είμαστε σε επαφή με τους σκιώδεις εισηγητές ε, για να σας φέρουμε έναν καλό συμβιβασμό που θα βοηθήσει όλους τους συναδέλφους που θέλουν να στηρίξουν τον προϋπολογισμό του 18 προϋπολογισμό ο οποίος θα μας δώσει μια ισχυρή θέση εν ώψη της συνδιαλλαγής και θα μας δώσει την δυνατότητα να υπερασπίσουμε τις πολιτικές προτεραιότητες για το επόμενο έτος που συναποφασίσαμε αρχές του έτους. Υπ' αυτήν την έννοια σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κύριε Μουρισάν. Άσβερ. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομο. Ε, θέλω να ευχαριστήσω του συνάδελφου για τα καλά του λόγια για την ε, δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Πολλά ε, πρέπει να γίνουν ακόμα. Αναμένω λοιπόν την περαιτέρω συνεργασία για να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα μπορέσουμε και εμείς να προτείνουμε να το πάμε στην συνδιαλλαγή με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου, Ρεσαν και Άσχουερθ. Τους ε, εύχομαι κουράγιο και φαντάζομαι ότι την Τυρκάς εβδομάδα θα την ευχαριστηθείτε όλοι, εκτός αν δουλεύσετε βέβαια, τέλος πάντων. Τώρα να περάσουμε στο πουδουπού για το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί από το 2021 και μετά. Χρειαζόμαστε τον εισηγητή μας, τον Γιάννη Ολμπεχτ και την εισηγήτριά μας, ε, την ε, Ιζαμπέλ Τομά, για να μας διαφωτίσουν και να ξεκαθαρίσουν το μυαλό μας το πώς έχουν τα πράγματα. Κυρία Τομά, ή μάλλον πρώτα, να πω ότι θα λήξει η συνεδρίαση 11 και 20 για να μπορέσετε να φτάσετε χωρίς να τρέχετε στην Ολομέλεια. Κυρία Τομά, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Άρα μου λέτε και εμένα να τρέξω τώρα ουσιαστικά. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως ξέρετε, αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε μετά από ε, το Reflection Paper Κρέτσου και ε, Έτιγκερ, να παρουσιάσουμε λοιπόν στο Κοινοβούλιο ένα ψήφισμα ως απάντηση σε αυτό το έγγραφο προβληματισμού. Το ψήφισμα προβλέπεται να ψηφιστεί τον Οκτώβριο. Όπως καταλαβαίνετε όμως, δεν θα έχει μπει σε μεγάλο βάθος γιατί χρειάζεται γι' αυτό η έκθεση πρωτοβουλίας που θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο για να ψηφιστεί το Μάρτιο. Για την έκθεση πρωτοβουλίας έχουμε ζητήσει από όλε τι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να γνωμοδοτήσουν για τις διάφορες πολιτικές που τις αφορούν. Είμαστε λοιπόν τώρα στη φάση που έχουμε ένα πολύ σύντομο ψήφισμα. Είναι μια πρώτη εκκίνηση, αν θέλετε, ε, για να συζητήσουμε τις γενικές κατευθύνσεις και τις προκλήσεις του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου για το μέλλον. Για το περιεχόμενο, γρήγορα-γρήγορα, να σας πω τι περιλαμβάνει αυτό το ψήφισμα. Πρώτα απ' όλα, Μιλούμε για το αόρια και τι ανεπάρκειες του τρέχοντος ποδοπού και του συστήματος χρηματοδότησης. Έπειτα χαιρετίζουμε το έγγραφο της Κομισιόν ως μέθοδο, αλλά λέμε ότι πρέπει να γίνουν διορθώσεις και να τροποποιηθεί το κείμενο πριν την ομιλία του Γιούγκερ. Βέβαια, έγινε αυτά γιατί υπάρχει μια φράση που λέει ότι το πέμπτο σενάριο είναι καλή, η αφετηρία και πρέπει να πάει πιο πέρα. Τώρα όμως έχουμε ένα άλλο σενάριο, το έκτο που μας παρουσίασε ο κύριος Γιούγκερ. Οπότε δεν πρέπει να είμαστε σε αντίφαση στο ψήφισμα αυτά τα οποία τελικά προβλέπονται. Επίσης, ότι αυτό το προηγούμενο πολιτές δημοσιονομικό ε, με βάση και την ανάλυση που είχαμε κάνει όλοι μαζί για την αναθεώρηση αυτού του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου και για τον Brexit λέμε ότι πρέπει το 1% του ΑΕΠ να πάψει να ισχύει ως όριο. Αυτό είναι το τρίτο. Και το τέταρτο, μιλάμε για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδιών πόρων ως κάτι απολύτως αναγκαίο με τη θέσπιση νέων ιδιών πόρων. Διότι σε διαφορετική περίπτωση θα ζητηθούν περαιτέρω εισφορές από τα κράτη-μέλη και αμφιβάλλουν για το κατά πόσο κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό. Επίσης επιλέγουμε μια, έναν ορισμό που θα περιλαμβάνει την έννοια της αξίας της Ένωσης και θέλουμε να υπάρχει μια πολλαπλή, πολυσχεδή ερμηνεία του όρου αυτού που δεν έχει οριστεί επαρκώ ακόμη. Επόμενο, ο προπολογισμό της Ένωση θα πρέπει να είναι βανάγνωστο και ευλήπτο για τους πολίτες, βασίζεται σε προτεραιότητε που είναι η βιώσιμη ανάπτυξη. Η αλληλεγγύη και η αμυντική ασφάλεια, ασφάλεια άμυνα κτλ θα πρέπει να τα βάλουμε όλα αυτά με τρόπο ορατό και εύληπτο. Επιμένουμε επίσης στην ανάγκη ο προεπολισμός να είναι ενιαίος και στην ανάγκη να προβλεφθούν μέσα που προς το παρόν εκτός προπλησμού, δηλαδή να ενταχθούν εκ νέου αυτά τα μέσα. Υπενθυμίζουμε στη συνέχεια ότι πρέπει να έχουμε ένα ευέλικτο δημοσιονομικό πλαίσιο για να μπορεί να προσαρμόζεται στις εξελίξεις, και επαναλαμβάνουμε τις προηγούμενε προτάσεις που είχαμε διατυπώσει στο πλαίσιο τη έκθεση πρωτοβουλία για την αναθεώρηση, δηλαδή πρόταση για το παθεματικό κρίση, επαναχρησιμοποίηση των ε, μη εκμεταλλευσών πιστώσεων και μιλάμε και για τις πληρωμές και τα ειδικά μέσα που πρέπει να είναι εκτό, του ορίου, του πλαφών για τα χρηματοδοτικά μέσα. Εκεί λέγονται διάφορα στον έγγραφο προγραμματισμού ε, την κύριε Κρέτσου. Λέμε ότι συμπληρωματικά τα εργαλεία δεν θα υποκαθιστούν τις επιχορηγήσεις, αλλά θα έρχονται συμπληρωματικά. Και αναφέρουμε τις ανησυχίες μας για την δένωση νέου ταμείου. Αν και θα ήμασταν έτοιμοι να εξετάσουμε το ενδεχόμενο δημιουργία ενό ταμείου εγγύσεων ενιαίου για τα δεματοδοτικά αυτά μέσα και ανησυχούμε για το αν θα ευθυγραμμιστεί ε, το χρονοδιάγραμμα με τις εκλογές για την Κομισιόν, για το Κοινοβούλιο. Ζητούμε τον αργότερο το Μάιο να καταθέσει προτάσεις της Κομισιόν για να μπορέσουμε εμείς να τις μελετήσουμε με ηρεμία, με ησυχία και να έχουμε και τις συζητήσεις μας με το Συμβούλιο διευκρινίζοντας ότι το Κοινοβούλιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκλειστεί αντίθετα να συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων. Merci, Ευχαριστούμε κύριε Ατόμα. Κύριε Όλμπριχτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να προσθέσω κάποια πράγματα σε αυτά τα οποία είπε η Τόμα, ότι η πρόθεση του ψηφίσματος ε, δεν είναι να καθορίσει το πεδίο εφαρμογή ε, συμφερόντων συμφερόντων του Κοινοβουλίου. Στόχος είναι η πολιτική θέση του Κοινοβουλίου. Πρέπει να πούμε λοιπόν ξεκάθαρα ναι και όχι. Αυτή είναι η πρόθεση. Οπότε, τώρα που είπαμε ε, ε, πρώτον αυτά τα κονδύλια δεν επαρκούν, ε, είναι σαφές. Και έχουμε λοιπόν ένα όχι για τα σενάρια αυτά. Γιατί δεν δεχόμαστε αυτό το οποίο είπε η Ιζαμπέλ Τωμά. Όχι για οροφή κάτω από 1%. Αντιθέτω, πρέπει να είναι πάνω από 1%. Ε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση να σπάσουμε το πλαφόν. Και κάτι άλλο το οποίο θέλω να επισημάνω. Λέει πως είτε θα έχουμε σύστημα ίδιων πόρων ή τα κράτη-μέλη πρέπει να δώσουν λεφτά. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Είναι ή όχι λοιπόν αν δεν βάλουν τους ίδιους πόρους δεν θα ε, υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει η δομή του προϋπολογισμού και είναι κάτι το πολύ συγκεκριμένο. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το στοιχείο ε, των πολύ διπλωματικών επιφυλάξεων για την πρόταση να μπουν μαζί όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που υπάρχει μες στο έγγραφο. και θα απαντήσουμε με τρόπο διπλωματικό. Κάτι άλλο για την διάρκεια. Ε, πρέπει να το δούμε στην Επιτροπή και της ε, Τροπολογής. Για τώρα λέμε 5 συν 5 ή 7. Γι' αυτό στο σχέδιο αυτό το οποίο θα τροποποιηθεί νομίζω πρέπει να ανοίξει αυτό για συζήτηση στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Γιατί ακόμα η συζήτηση συνεχίζεται. Αυτή είναι η προσωπική μου παρατήρηση που δεν θα τη συζητήσουμε ότι πρέπει να ξέρουμε πριν οριστικοποιηθεί αυτό το έγγραφο τι σημαίνει, τι σημαίνει η νέα γραμμή υπερπολογισμού για την Ευρωζώνη. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο συνέβη χτες και ο δικός χάρτης λέει ότι η πρόταση για τη νέα γραμμή προπολογισμού για την Ευρωζώνη θα είναι έτοιμη τον Δεκέμβριο φέτος η πρόταση. Τι σημαίνει αυτό για το ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ εντάξει να προσθέσουμε κάτι, αλλά είναι μια ιδέα ή είναι θέμα νέων κονδυλίων, φρέσκων κονδυλίων, τι είναι. Τι σημαίνει νέα γραμμή υπερπολογισμού για την Ευρωζώνη. Για να συνοψίσω. Δεν θέλουμε απλά ένα άλλο νέο έγγραφο που λέει καλύτερα υγι... νέος και υγιής και πλούσιος παρά ε, γέρος και ασθενής και φτωχός. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ολμπριχτ, ευχαριστώ και τους δύο συγγητές μας. οι οποίοι εξερευνούν ένα πεδίο του προπολογισμού το οποίο ενέχει πολλές ε, βεβαιότητες. Διότι στο Πουδουπού 2014-2020 με την κρίση δεν τα καταφέραμε όλα, δεν τα λάβαμε όλα υπόψη. Οπότε είναι σαν να προσπαθούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα ποια θα είναι η Ευρώπη σε λίγα χρόνια. Τι αρμοδιότητες θα πρέπει να εξασκήσουμε και να προβλέψουμε για να είμαστε αποτελεσματικοί δουλειά και το καθήκον της Ιζαμπέλ και του Τάς έχουν γίνει ιδιαίτερα δυσκερείς. Θα ζητήσω από τους σκιώδεις μας να μας πούν την άποψή τους, ο κύριος Κέλμελ πρώτος. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ ιδιαίτερο τους δύο συνεισηγητές για την δουλειά που έχουν κάνει και θα ήθελα εγώ να αναφέρω μια εσωτερική αντίφαση που υπάρχει. Αφενός ε, αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να αποφασίσουμε τώρα τι μορφή θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Ε, τα είπε και ο Ζαν Κλοντ ε, χτες, ποιο είναι το όραμά του αλλά λέμε ότι βεβαίως πρέπει να περιλάβουμε και τους ε, πολίτες. Αλλά όταν ταυτόχρονα λέμε ότι αυτά τα πράγματα δεν τα αμφισβητούμε καθόλου, δεν ξέρω. Νομίζω ότι καθορίζουμε από τώρα πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να καθορίσουμε γιατί πολλοί από εμάς ε, λέμε ότι πάντα πρέπει να προχωράμε παραπέρα, να έχουμε όλο και περισσότερα, αλλά γνωρίζουμε ότι πολλοί πολίτες δεν το θέλουν αυτό το πράγμα. Και να λέμε μόνο το τι αρμοδιότητες έχουμε και ότι θέμε λεφτά, δεν φτάνει. Αποφασιστικό είναι και το ερώτημα ποιος πρέπει να ασκεί αυτές τις αρμοδιότητες αν πρέπει να τις ασκεί όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση ή μήπως αποτελεσματικότερα μπορούν να ασκηθούν από τα κράτη-μέλη. Και αν καταλήξουμε στο αποτέλεσμα ότι χρειάζεται λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις αρμοδιότητές της, πρέπει πάντα να πούμε ποιος πληρώνει. Υπάρχει ε, διάθεση για κάτι τέτοιο, γιατί γνωρίζουμε πως πολλά κράτη-μέλη δεν είναι διατεθειμένα να πληρώσουν ε, περισσότερο. Όλοι θέλουν περισσότερα από όλου, αλλά πρέπει να ρωτηθούμε σε ποιου τομεί θα οι πολίτες μας να έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο δεν το έχουμε ρυθμίσει αυτό, δεν μπορούμε να καθορίσουμε τίποτα. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει πρώτα με τους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη και μετά να βρούμε τις διάφορες εναλλακτικέ που υπάρχουν και πάντα να λέμε πόσο κοστίζει. Αυτό πρέπει να κάνουμε νομίζω συνολικά και καλό θα ήταν να μην έχουμε πάντα έτοιμη την κατανομή και να λέμε ότι κάποιοι είναι υποτίθεται φίλοι της Ένωσης και κάποιοι εχθροί της Ένωσης ε, υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι υπάρχουν άλλε καλύτερε λύσεις. Αυτό δεν σημαίνει εχθρός της Ένωσης, σημαίνει εχθρός της αναποτελεσματικής Ένωσης και των παράλογων λύσεων. Γιατί εγώ αισθάνομαι ότι αυτή είναι η υποχρέωσή μου απέναντι στους φορολογούμενους της Ευρωπαϊκής Ένωση. Όχι, όχι. Δεν υποπτευόμεθα εσάς, κυρία ο κύριος Σολέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση για το πολιετές το επόμενο σίγουρα είναι μια από τις σημαντικότερες συζητήσεις για τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Γιατί για τις πολιτικές χρειάζονται λεφτά και με τον προπολογισμό φαίνεται αν έχουμε πραγματικά ε, την απαιτούμενη προσήλωση ή όχι για την επίτευξη των στόχων. Φυσικά, η συζήτηση για το νέο πουδουπού έχει άμεση σχέση με τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Τι είδου Ευρώπη θέλουμε για το μέλλον. Άρα, ο προπολογισμό πρέπει να αντικατοπτρίζει και την ιδέα που έχουμε για την Ευρώπη. Και εγώ προσωπικά προσωπική παρατήρηση, θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο ισχυρή, με περισσότερες αρμοδιότητες και πιο ικανή να αντιμετωπίσει τις ανάγκες και να ικανοποιήσει τις επιθυμίες των πολιτών. Το έγγραφο της Κομισιόν είναι μια καλή βάση συζήτηση. Είναι καλό έγγραφο κατά την άποψή μου. Έχει κάποιες καλές ιδέες. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές για το έργο τους, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Με την πρόταση ψηφίσματος. Δύο δέσμες προβλημάτων θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο προσεχές ε, πουδουπού. Ποσοτικά επιχειρήματα φενός και ποιοτικά επιχειρήματα φετέρου. Σε ό,τι αφορά την ποσοτική Πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία για το συνολικό ύψος. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει από το 2020 να μειωθεί το επίπεδο των πόρων. Και επίσης θα πρέπει να δούμε τη δομή των εσόδων και να την αναθεωρήσουμε πλήρως. Να έχουμε δηλαδή ένα προπολογισμό χωρίς καμία έκπτωση και επιστροφή και να χρησιμοποιούνται μόνο οι διπόροι, στο κατά κύριο λόγο για τη χρηματοδότηση του προπολογισμού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά θέματα, θα πρέπει να δούμε τι προτεραιότητες θέλουμε να εφαρμόσουμε με τα χρήματα του προπολογισμού. Κοινωνικέ ανάγκε, ε, ευάλωτοι πολίτε, εδαφικές ανισότητες, ο προπολογισμό πρέπει να υποστηρίξει μια ανθεκτική ε, προσανατολισμένη προ το μέλλον οικονομία. Θέλουμε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο που θα αντιμετωπίζει την αλλαγή του κλίματο. Άρα, πιο πράσινο προπολογισμό. και πολιτικέ κατά τη κλιματική αλλαγή. Θέλουμε τέλος έναν πιο διαφανή προπολογισμό με έλεγχο, να μπορούν οι πολίτες να ελέγχουν τον πολιτισμό αυτό περισσότερο από ότι τώρα. Αυτά είναι κάποια από τα πιο σημαντικά θέματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σολέ. Κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Ουδής. Αν με επιτρέπετε δύο λέξεις. Το σημαντικότερο είναι πράγματι να αρχίζουμε να οραματιζόμαστε την αυριανή Ευρώπη. Υπάρχει παγκοσμιοποίηση και σε ό,τι αφορά προνόμια εθνικής κυριαρχίας, τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να έχουν αυτή την εθνική κυριαρχία. Στο ψηφιακό επίπεδο, για παράδειγμα. Πολυεθνικές δεν δίνουν καν φόρο, το ΙΚΑΦΑ, οι τέσσερις αυτές ε, πολυεθνικές. Δεν δίνουν πλέον τους φόρους τους. Και επειδή είπαμε για αμυντική βιομηχανία, εξοπλισμούς και έχουν και την καταπολέμηση δημοκρατίας, έχουν πρόβλημα μετανάστευσης. Ίσως πρέπει κάπως να στερέψουν οι πηγές τη μετανάστευσης. Έχουμε 800 εκατομμύρια Αφρικανών ε, ε, τις επόμενες χρονιές που θα έρθουν εδώ, αν ζουν ακόμα. Τι αλληλεγγύη θέλουμε και πόσο αποτελεσματική θα είναι μια Ευρώπη που θα μας προστατεύει. Γιατί αυτό ζήτησε ο Γιούνκερ, ότι θέλουμε μια Ευρώπη που να μας προστατεύει και που θα καλύψει το δημοκρατικό της έλλειμμα. Γιατί σήμερα δυσκολεύεται να μιλήσει πολύ της Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για τους ίδιους πόρους. Δεν είμαι σίγουρος ότι οι ίδιοι πόροι σημαίνουν συμπληρωματικοί πόροι, πρόσθετοι πόροι. Απλά η δίκαιη επιστροφή ως έννοια ε, καταργείται. Υπό την έννοια ότι δεν βάζουν το χέρι στην τσέπη τα κράτη και μετά να υπολογίζουν τι πήρα και τι έδωσα. Πρέπει να ορίσουμε τους ίδιους πόρους, πρέπει να τους ορίσουμε ξεκάθαρα. Αν είναι δημοσιονομικού χαρακτήρα, φορολογικού χαρακτήρα, θα έρθουν να προσθεθούν στους εθνικούς και τοπικούς φόρους αλλά δεν θέλουμε να συνθλίψουμε τους φορολογουμένους. Πρέπει να υπάρχει πόνο λοιπόν στο αντιστάθμισμα ελάφρυνση των εθνικών φόρων. Είναι ήδη όμως 11 και 20. Παραμίλησα. Αλλά πρέπει να ακούσουμε και ε, τον Επιτροποτές πάντων. Πότε πρέπει να ψηφίσουμε. Πριν το 19 τις εκλογές. Θα αφήσω τον τελευταίο λόγο στους συγητές. Ποιος από τους δυο σας θέλει να πάρει πρώτα το λόγο, ο κύριος Όλμπριχτ. Μια παρατήρηση. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Κέλμε. Δεν είπα αυτό που λέτε. Συμφωνώ με τη μεθοδολογία. Έτσι ακριβώς πρέπει να είναι. Η συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Και το δεύτερο, οι αρμοδιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λέμε οι περισσότερε, όχι λιγότερε εκεί διαφωνώ. Αυτό είναι το δεύτερο. Και τρίτο βήμα. Πόσο θα κοστίσει. Τέταρτο βήμα. Με τι μέσα. Δεν δουλεύει όμω, Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι ο ιδανικό κόσμο που δεν υπάρχει όμω. Εμεί θα πρέπει να απαντήσουμε ω Επιτροπή Προπολογισμών τα ερωτήματα που δεν θα θέσουν οι άλλοι. Περιμένουμε από το Συμβούλιο να λάβει την απόφαση τι πρέπει να είναι στο μέλλον Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά ποιες επιπτώσεις θα έχει αυτό στον προπολογισμό. Εμείς θα κάνουμε ε, το μοντέλο από τον προπολογισμό και όχι το ανάποδο. Δεν ζούμε σε έναν ιδεώδη κόσμο. Δηλαδή μπορεί να διαφοροποιούμαστε στο το περιεχόμενο, αλλά συμφωνώ ότι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τι να κάνουμε. Και άτομα παντώντα στα ερωτήματα που ετέθησαν, πρώτα απ' όλα το Συμβουλίο είπε πως ορίζει το μέλλον της Ευρώπης, αλλά το ίδιο έχει κάνει και το Κοινοβούλιο. Και εμείς έχουμε δικαίωμα να μιλάμε και να λέμε τι πιστεύουμε για τις αρμοδιότητες που θα πρέπει να έχει ή δεν θα πρέπει να έχει ένωση. Τούτου λεχθέντος. Υπάρχουν αρκετά ερωτήματα. Πρώτον, έσοδα και, δημοσιο... και δομή του προπολογισμού. Εκ την έκθεση πρωτοβουλία για το μελλοντικό ποδού, που υπάρχει και μια άλλη έκθεση που θα ψηφιστεί ταυτόχρονα για τους ίδιου πόρους. Άρα έχουμε να βάλουμε τα πόδια μας και στις δύο βάρκες και να πηγαίνουμε ταυτόχρονα. Για να απαντήσω στον κύριο Σολέ. Για το περιεχόμενο δεν έχουμε αρχίσει να συζητάμε ακόμα. Και στον κύριο Κάλμελ απαντάω ταυτόχρονα. Γιατί περιμένουμε το input από τις επιτροπές. Εμείς ως Επιτροπή Περιπολογισμών δεν είμαστε παντοδύναμες για να αποφασίσουμε Θέλουμε να δούμε, θα μας πούν και άλλες επιτροπές. Τρίτον, έχουμε κάτι καινούριο. Μετά την ομιλία του Γιούνκερ χθε, γιατί το draft το είχαμε ετοιμάσει πριν την ομιλία του Γιούνκερ, αλλάζουν τώρα τα πράγματα. Και υπάρχουν και πολλά θέματα που θα πρέπει να αναφέρουμε. Ίσως όχι στο ψήφισμα βέβαια. Μάλλον στην πρωτοβουλίες. πρωτοβουλία. Που την έχουμε λίγο βάλει κατά μέρο πώ το Μίλησε τη διάρκεια κ. Σόλμπριχτ, αλλά υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Οι όροι, οι προποθέσει. Αυτά τα ανέφερε χθε ο Ζαν Κλοντ Ιουνκέρ. Και εμεί θα πρέπει να τα συζητήσουμε και θα έχουμε μια πολύ έντονη συζήτηση για τι πολιτικέ ελευθερίε, για τη μακροαρεσιμότητα, για του μετανάστε. Ξεκάθαρα άφησε ο Γιούνκερ αυτά τα θέματα. Θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση και τι θα γίνει με, το, με την Ευρωζώνη και την ουσιανική κάτω. Και αυτό πρέπει να το πούμε και αν τα δούμε. Μπορεί να αποφύγουμε να αναφέρουμε την επιθέματα τώρα στο ψήφισμα, αλλά δεν μπορούμε να, συστή, να μην τα αναφέρουμε στη συνέκτηση τη πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε. Πρέπει ο προπολογισμό να συνοδεύεται από πολιτική θεώρηση και βούληση. Και όταν λέω θεώρηση, ελπίζω ότι ο προπολογισμό ανταποκρίνεται στι πολιτικέ μα φιλοδοξίε και ότι το χάσμα αυτό δημοκρατία θα καλυφθεί σύντομα από γέφυρε με μια σύμβαση για την Ευρώπη. Η σύμβαση των πολιτών, η συνέλευση. Επόμενη συνεδρίαση 26-27 Σεπτεμβρίου. Άκρο σημαντική, διότι θα ψηφίσουμε τι τροπολογίε και τι συμβαστικέ για τον προπολογισμό το 2018 και θα είναι και η ευκαιρία μας να εξετάσουμε τα άλλα ζητήματα που ήταν σήμερα στην ημερήσια διάταξη αλλά για λόγους χρόνου δεν μπορέσαμε να τα καλύψουμε. Ε, λίγη συνεδρίαση.